Imod? Hverken eller. Det kontrollerer vi. Der stemmes om 68. And it's closed. Έκλεισε η ψηφορία. Δεκτή 69 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή τι η 70 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 109 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.39 υπέρ κατά 3. Λυπάμαι, έκανα λάθος. Απορρίφθηκε η συμβαστική πρόταση. Έτσι, λυπάμαι λοιπόν ε, ψηφίζουμε για την 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα ψηφίζουμε για το 239. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 240. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 241. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές 74 και πάλι υπέρ κατά αποχές, συγγνώμη, ηλεκτρονική επαλήθευση. Και για μένα είναι καινούργια η διάταξη, δεν είναι η συνηθισμένη αίθουσα που ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα παρακαλώ και έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται, δεκτή η τροπολογία. 2.42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 όχι καταπίπτει η 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στην ε, συμβαστική 15. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβαστική 15. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται δεκτή η συμβαστική. Συμβαστική 16. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 17 έκλειση ψηφοφορία δεκτή η τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται συγγνώμη 114 υπέρ κατά αποχές ε, ε δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. 120 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. 123 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή είπα 125 αλλά κανονικά ήταν ένα μπλοκ τροπολογιών μέχρι την 131 Τώρα πάμε στην 136 πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 19. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή. απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Μισό λεπτό. Ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα μοιάζαν πάρα πολύ. 155 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2. Κάτι έχω χάσει κάτι. Πάμε στη σελίδα 14. Προχωρήσαμε πάρα πολύ. Η 15 ψηφίσαμε για την ε, ε τροπολογία 1 και τώρα ψηφίζουμε για την 2 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 λέει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές δεκ... απορρίπτεται. 208. Πάλι το ίδιο λάθο έκανα, λέει η πρόεδρο. Τροπολογία, συγγνώμη, συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 206. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 207. Υπέρ, κατά, αποχε εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. 2.10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.12 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 2.12. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Αποτέλεσμα δεκτή. Συμβεστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Πάλι έκανα λάθος. Έχουν πάλι εδώ κάποια χρώματα και μπερδεύομαι. 2.15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, ε, δεκτή. 2.18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 ε, τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 18 η καταπίπτη 18 όπως και η 19 πάμε στην 20 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 ε, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η 225 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Όχι, πίπτη. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 37 καταπίπτει. Η 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. Η 2.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 2.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, την τελική. Μπορείτε να ψηφίσετε. Closed. Πέρασε. Και εγκρίθηκε. Now we vote. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία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 Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Και η πράσινη ήταν ε, κατά. Α, πρόσεχα πως ψήφισε η άλλη και δεν το πρόσεξε. Ωραία, τροπολογία 3 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές Δεν ξέρω. Για την 4. Ποιος είναι υπέρ. Ωραία, εγκρίνατε τότε. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ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 Πέρας της Εγκρίθηκε με ομοφωνία. 67 ψήφισαν 67 υπέρ. Εγκρίθηκε λοιπόν. Και τώρα περνάμε στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές της ε, σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ψηφίζουμε σχέδιο γνωμοδότησης. Και αρχίζουμε με την τροπολογία αριθμός 31. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για την 89 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της προφορίας. Εγκρίθηκε. Να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ στην ψηφοφορία για να μην κάνω τέτοια λάθη. Να βλέπω τα χέρια σας. Για μένα ήταν προφανές ότι είχε απορριφθεί. Λοιπόν, 85 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Ωραία. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Στην τροπολογία 94 της κυρίας Κοτνέτσα πάλι, οπότε να βλέπω τα χέρια σας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δέκα, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας εγκρίθηκε. Καταπίπτουν επόμενες. 99 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεκατέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεκαπέντε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά. Βλέπω πολλά χέρια να σκόνται κατά, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 113. Δεν καταλαβαίνω πώς ψηφίζουν οι ομάδες. Ποια ομάδα ψηφίζει πώς. 113 λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 117. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. 119 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε για την 119. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίζετε. Πέρας της φοφορίες. Απορρίφθηκε. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 και 131 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 132 και 133 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 134-135 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 136-137 υπέρ, όχι, Α, καταπίπτει αυτή. Περνάμε στο 17. Από ό,τι φαίνεται καταπίπτει. 17 υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε. Close. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη σελίδα, του 140. 140 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 146-151 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 149-155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 153 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 154 υπέρ, καταπίπτει, 154, α, αυτό κοίταζα και είπα 5, υπέρ του 154, κατά αποχές εγκρίνεται, 156 υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε το 160 ψηφίζουμε για την 160 πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 162 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το 164. Κυρία Γκαρντίνη, τι ψηφίσατε. Στο 164 ήταν ε, συν 32 μείον 33. Ε, είναι σημαντικό, ναι, και είναι λάθος. Εγκρίνεται, λοιπόν.

τώρα πήραν μέρος σε περισσότερη ψηφοφορία από ό,τι πριν. Α, 165 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 166 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 167 υπέρ, κατά, αποχές, για να ελέγξουμε για το, 167. Η Μαριάννα που είναι. Πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται. Είμαστε στο 168, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 170 υπέρ. Κατά αποχές, για να ελέγξουμε. Πέρας ναι, ψηφοφορία. 171 ναι. ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε για την 174. Ε, Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 173-175 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 καταπίπτει. Περνάμε τώρα στο, την 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε. Καθυστερήσατε να σηκώσετε το χέρι σας. Ωραία, απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε για να ελέγξουμε πάλι το 187 την 187 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 και 92 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 α μισό λεπτό να ελέγξουμε το 195 Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 199 είναι ταυτόσιμη. Περνάμε τώρα στο 200. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 υπέρ, ε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, για να το ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το, θα πρέπει το FTD και η ΜΕΒ να σηκώνουν τα χέρια τους και στην ΚΟΕ γιατί στις τελευταίες ψηφοφορίες δεν ήταν ξεκάθαρο τι θέλετε να ψηφίσετε. Περνάμε τώρα στο 206. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για να ελέγξουμε. Και πάλι, και πάλι δεν βλέπω τα χέρια σας. Κυριεύει. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 216 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε το 2, την 216. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 2.14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.18 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 2.19. Υπέρ. Α, καταπίπτει. 2.21. Υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Πέρας πληροφορία. Εγκρίνεται. 2.22. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.30 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε την 2.31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.32. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.33. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, για να ελέγξουμε την 27. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές Για να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.51 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ 32 υπέρ κατά, υπέρ... Α, μισό λεπτό. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε. 39. Άρχη ε, ψηφοφορία, ε, ψηφοφορίας, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40. Ψήφι Κατά. Για να ελέγξουμε για το, την 40. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 42. Υπέρ, κατά, αποτιές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε την ε, τροπολογία 1. Αρχι, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο ε, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά Την 46 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 53 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 54 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 56 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές για να ελέγξουμε την 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνηκε. 57. Όχι, περάμε στις 5. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 5. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε πάλι. Ε, ε, ε, πέρας, δεν λειτουργήσαν εδώ οι συνήθεις συμμαχίες, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ψηφίζουμε για την 6 αρχή της ψηφοφορίας Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 74. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά. Για να ελέγξουμε την 80, η ηλεκτρονική ψηφοφορία την 80. Πέρες ψηφοφορίας απορρίπτεται. 81. Η ψήφι υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. So, we come to the main attraction of this evening. Ε, στο τελικό, πιο σημαντική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για τα αυτοκίνητα. Πρόκειται για τις, ε, ε, λεπτό, πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια λαφρά επαγγελματικά οχήματα. Αναδιατύπωση. Ε, να έχετε λίγο υπομονή, ε, γιατί θα πρέπει να κάνουμε πολλές επαληθεύσεις και να σηκώνετε τα χέρια σας. Συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ. Συμβαστική 1. Εγκρίνεται. Πολύ καλή αρχή. Συμβαστική 6α. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 6α, παρακαλώ. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, περισσεύουν δύο. Τώρα περισσεύει ένας. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Συμβαστική 6β καταπίπτει. Συμβαστική 7. 7. Ας ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την ε, συμβαστική 7. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. Η 13. Πάμε στην 8α. Και πάλι λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι 8β καταπίπτει. Η 277 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Τραν 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. Η 280 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 296 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Είσαστε κατά. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε. Για αυτό το μπλοκ, ποιος είναι παρακαλώ υπέρ. Κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Και έκλεισε η ψηφοφορία και γκρίνεται. Τραν 38 και 50. Για αυτά τα δύο μπλοκ ψηφίζουμε, παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,97 και τραν 39. Ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε 3.15 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται. 3.18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.19 και 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 322 ε, με 325 και τραν 42 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Και έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Η 330 και 172 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 326 μέχρι 329 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 43 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.32 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση 3.32. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και γκρίνεται. Τραν 44 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 333 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 334 και 335 υπέρ παρακαλώ και η 33. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 και τραν 5 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Η τραν 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 345 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υπέρ, κατά, όχι καταπίπτει. Επειδή κατέπεσε η 3.45, καταπίπτει και η 112. 3.41. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.42. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.43 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 3.44 υπέρ κατά αποχές 3.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 347-349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 350 και 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 348 ψηφίσαμε για αυτήν. Η 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11α, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. με μία ψήφο διαφορά, όχι δύο. Η 11 β συμβαστική υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 11 β. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία και απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για τις τροπολογίες υπό την συμβιβαστική. Ξεκινάμε με τη 281 και την 164. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 37, 372, 373. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για αυτήν παρακαλώ. Ψηφίζουμε. και έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 166 ψηφίζουμε παρακαλώ. και η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Η 17 υπέρ καταπίπτει. Α, κατέπεσε η 17 Θα προχωρήσουμε τώρα λιγάκι γιατί κατέπεσε η 166 Πάμε στην 374. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Η 374. Και πάλι. Υπέρ. Υπέρ της 374. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήτευση. Ψηφίζουμε. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, γιατί είναι, πρόκειται περί συμβαστικής πρότασης. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Και κλείσει η ψηφοφορία. Και γκρίνεται. Τροπολογία 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ξεκινάμε με την 30 και πάει μέχρι το 4.15. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιατί 406 ήταν αυτό. Και πολλές καταπίπτουν ε, τι απορρίφθηκε το 8, απορρίπτεται 406, πάμε στην 407, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 411, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 416 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα μισό 360 Τρία εξήντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Συμβαστική 2α. Ψηφίζουμε παρακαλώ. και έκλεισε και απορρίφθηκε. Η 2β ηλεκτρονικά Ψηφίζουμε τώρα για την 2β. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Άρα θα ψηφίσουμε για όλες τις τροπολογίες. 419 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 420 και 184 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. 421 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 422 και οι 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 48 και 21 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. 48-21 υπέρ έκλειση ψηφοφορία απορρίπτεται. Τραμπ 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 426 υπέρ ε, από κοινού με την 535 και 654 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 423 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 423 ψηφίζουμε παρακαλώ απορρίφθηκε 424 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τραν 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 49. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 4.29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 και η 436 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για αυτήν. Ψηφίζουμε. Και έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. 4.35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία, απορρίπτηκε. 442, 443 μπλοκ υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και γκρίνεται. 444 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Λοιπόν, προχωράμε τώρα λίγες σελίδες. Ψηφίζουμε για ένα μπλοκ για την 55, 468 και 469, αλλά μάλλον καταπίπτουν και αυτές. Όχι, αυτές καταπίπτουν. Α, προχωράμε πολύ. Μπράβο. Μου λέτε λιγάκι που πάμε. τα δικά μας χαρτιά 529, σελίδα 53, 529 παρακαλώ. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της 529. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. και κλείσει ψηφοφορία και απορρίπτεται. Σελίδα 55 η 539 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική παλίτεψη, Και έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Σελίδα 58 καταπίπτει. Γιατί μου λέτε. You mentioned... Είμαστε στην τροπολογία 58. Σελίδα... Okay. Ήταν μετά είναι η Τραν 73. Ποιοι υπέρ. Κανείς. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 78. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Τραν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίθηκε. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 6 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τραν 8 και 9 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 89. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Εκατόν τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, 101 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τραν 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω να θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για την Τραν 13. Ψηφίστε. Θα άλλαζε αν εγκρίναμε κάτι από την Τραν. Τέλος. Εγκρίθηκε και όμως. Ωραία. Συνεχίζουμε και πάμε στη συμβιβαστική 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ. Α, καταπίπτει. Δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Όχι. Πάμε στη σελίδα 78. 131. Πρέπει να ψηφίσουμε 131 πρώτα. Υπέρ. Κατά. 131, έτσι. Στη σελίδα 77. Υπέρ, παρακαλώ, της 131. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 141 τώρα. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 141. Τέλος. Απορρίφθηκε. 15. Α, καταπίπτει 15. 152 τώρα, στη σελίδα 79. 152 δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 321 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 157 μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τραν 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 175. Ψηφίστε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Και τώρα προχωράμε και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ή έχουμε κάτι ακόμα να ψηφίσουμε. Αν δεν έχετε αντίρρηση, περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, έτσι, τελική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε.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 Τώρα, ψηφίζουμε για την ποιότητα του νερού προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, επαναδιατύπωση. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης. Τροπολογία 118. 118, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. Ωραία. Θα ελέγξουμε γιατί είναι συμβαστική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. 1Β. Πέρα στις ψηφοφορίες και απορρίφθηκε. Συμβαστική 1α ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. «296 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά». 296. Τέλος. Απορρίφθηκε. 297 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 298 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 304 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 306 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 307 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 308 και 309 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ, κατά, αποχές, τελέξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 324 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 346 και 347 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, να ελέγξουμε. Καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 372 υπέρ. «369 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 372 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ε, ε, ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 401 υπέρ κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 402 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 403 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 20. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19α υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 19β τώρα υπέρ. Ηλεκτρονικά, έτσι καλύτερα. 19 Β. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 19 Σ. Υπέρ. Α, ηλεκτρονικά είπαμε. Ναι, σωστά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. 19 Σ. Εγκρίθηκε. Οπότε, φτάνουμε συμβαστική 12 και συμβαστική 22α μαζί. Συμβαστική 12 με τη συμβαστική 22β τώρα. Ηλεκτρονικά καλύτερα, γιατί είναι συμβαστική. Ψηφίστε. 12 και 22 β. Αυτό ψηφίζουμε. Όχι το α, το β, 22 β Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. «465 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 466 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 466. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 467. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε. Εγκρίθηκε η 15α, ε, 15α ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Σελίδα 34. Συμβαστική 16. Α, μισό λεπτό. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, 669 και 670 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 672 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 673 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα 674 και 675 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 676 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 682 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 683 και 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 685 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 685 ηλεκτρονική επαλήθευση και κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται τώρα ψηφίζουμε γιατί την 686 και 687 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 688 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή ε, ας κάνουμε ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 688. Ψηφίζουμε παρακαλώ και η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 689. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 690. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση 690. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε απορρίπτεται. 691 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 692 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 693 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 694 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 695 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 696 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε παρακαλώ και έκλεισε η ψηφοφορία και γκρίνεται 697 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ καταπίπτει Λοιπόν, καλό, ωραίος αριθμός, αλλά δεν ψηφίζουμε γι' αυτόν. Προχωράμε. 700 ή 700 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 701 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. 702 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 και 704 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 703 όχι κατέπεσε Πάμε στα παραρτήματα. Ε, συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 732 υπέρ κατά αποχές ε, είναι κανείς υπέρ Έκλεισε η ψηφορία. απορριπτεται Απορρίπτεται. 3-3. Ε, who is in favor? Against. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 743 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 744 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. απορρίπτει. αποχές απορρίπτεται. 746 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 747 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας, ψηφίσουμε για την 747. Πέρας ψηφοφορίας. Όλοι ψηφίσατε θετικά. Εγκρίνεται. 748. 748. Η ψήφη υπέρ, κατά, αποχές. Η πράσινη Ωραία, για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τουλάχιστον τρεις ομάδες δεν ψήφισαν κάτι. Πέρας ψηφοφορία, εγκρίνεται. 749 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 750 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 751 ψήφι πέρα. Κατά αποχές απορρίπτεται. 109 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 752 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 753 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 754 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 755-756 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 25. Ψήφι υπέρ, κατά. Ε, το ελέγχω ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τις τροπολογίες 772 μέχρι 74 ψήφι υπέρ των τριών τροπολογιών. Κατά αποχές απορρίπτεται 781 υπέρ καταπίπτει. Καταπίπτει. 786, 787 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 52. Ψηφίζουμε την τροπολογία 822. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 849 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Για να κάνουμε ένα έλεγχο ηλεκτρονικό, ελέγχουμε την τροπολογία 849. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 850 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Από ό,τι φαίνεται ψηφίζουμε τη συμβαστική πρόταση 26α. Συμβαστική πρόταση 26α. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. 26α. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27. Συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1.24, ψήφι υπέρ, <coughs> κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε. 124. Πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. 125 ψήφι πέρα κατά αποχές απορρίπτεται, 126 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 127 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ο κύριος Γεργάντη. Α, κύριε Γεργάντη, δεν με βοηθάτε αφού δεν σηκώνετε το χέρι σας. Πέρα της ψηφοφορίας. Ή μάλλον ε, δεν βοηθάτε την ομάδα, γιατί δεν ε, ε, χρειάζεται να κάνω ηλεκτρονικούς ελέγχου συνέχεια. 128 ψήφι υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε πάλι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 129. Ποιος είναι υπέρ της 129. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική πρόταση 30 ή 30 καταπίπτει Α, δεν εγκρίνεται η 19.1, Συνεπώ καταπίπτει αυτή η συμβαστική πρόταση και περνάμε σε μονομόνες ε, τροπολογίες. Ξεκινάμε με την 140, υπέρ, κατά, 140, ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 142, υπέρ, είναι ταυτόσιμη. 141, Καταπίπτει. Είναι ίδια. Ωραία. Περνάμε στις 146, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 31 καταπίπτει, ψηφίζουμε ξεχωριστά, 148 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και 152 ψήφι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 32 συμβιβαστική πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά μια ελέγξη ελέγξουμε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά υπέρ κατά 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές ε, για να την ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 37 υπέρ κατά, ε, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 192 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική πρόταση 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 196 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε, για να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 196. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 39, ψήφι υπέρ. Περάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 199 ψήφι ΠΕΡ, ψήφι κατά, απορρίπτεται. Η Συμβαστική Πρόταση 14, υπέρ κατά εγκρίνεται. 208 ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 41 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2.14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2.13 υπέρ α καταπίπτει. Συγγνώμη λέει πρόεδρος. 215 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ Ένα πρόβλημα με τον ήχο υπήρξε και δεν ακουγόταν η πρόεδρος στην καμπίνα καθόλου. 236 τώρα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 237 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. 19 με 41 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 242 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 45 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 247 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 249 επέρ. κατά, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Αυτή ήταν η τελευταία μας ε, ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και θα τα πούμε την Πέμπτη. Στο μεταξύ βέβαια και στην Ολομέλεια. Καλό βράδυ σε όλους.